Ο κύριος Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να καθίστε για να αρχίσουν οι ψηφοφορίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ. Πρόκειται να αρχίσουν οι ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσουμε με ονομαστική ψηφοφορία, η οποία έχει ζητηθεί. Καθίστε λοιπόν. Η κυρία Φρασόνη επί της διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε, Μία μικρή παρέμβαση, γιατί οι συνάδελφοι δεν έχουν ακόμα καθίσει όλοι. Αλλάξαμε τον κανονισμό γιατί περνούσαμε πάρα πολύ χρόνο σε ανώφελες συζητήσεις και αποφασίσαμε ότι σε ό,τι αφορά την έκθεση Άουκεν δεν θα διεξαχθεί συζήτηση.